Έχω να σας πω τα εξή σε σχέση με την ε, επανάληψη της Συνόδου. Αυτή τη στιγμή ε, ασχολούμαστε με τους νότιους γειτονές μας. Πρόσφατα Έπνευσαν νέοι άνεμοι στην Αίγυπτο και θαυμάζουμε την παρησία του Αιγυπτιακού λαού που επέφερε σημαντικές αλλαγέ στη χώρα, αλλαγέ τι οποίες υποστηρίζουμε. Λυπούμεθα για την απώλεια ανθρώπινων ζωών φυσικά και καλούμε όλες τις κυβερνήσεις των, ε, της περιοχής να έλθουν σε διάλογο με τους πολίτες, ε, να μην γίνονται διώξεις ε, των διαδηλωτών που διαδηλώνουν ειρηνικά και όπου επικρατεί στρατιωτική κατάσταση εδώ και χρόνια θα πρέπει να ακουστεί πια η φωνή του λαού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ε, καθήκον για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για καθέναν από εμά. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το 1989 πολλοί ε, Ευρωπαίοι πολιτικοί ανησυχούσαν για τις αλλαγέ που είχαν ε, δρομολογηθεί στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Α μην φοβόμαστε να εμπλακούμε πολιτικά και οικονομικά. Α βοηθήσουμε τους γειτονέ μας που έχουν δημοκρατικέ φιλοδοξίε, α του βοηθήσουμε να ζήσουν αξιοπρεπή ζωή στι χώρε του. Α μην του εξαναγκάσουμε να μεταναστεύσουν,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 σε σχέση με τα γεγονότα στις ε, νότιες χώρες, ε, γείτονες χώρες, να σας πω ότι ευρωπαϊκές χώρες, ε, πολλές ευρωπαϊκές χώρες δέχονται μεγάλο αριθμό μεταναστών από τις εν λόγω χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενεργήσει ταχύτατα και να υποστηρίξει τις χώρες αυτές που αντιμετωπίζουν μεγάλη ζωή προσφύγων. Και αυτό είναι καθήκον όλων μας, είναι μια κοινή ευθύνη. Στις 12 Φεβρουαρίου ήταν η Διεθνής Μέρα κατά των ε, παιδιών ε, στρατιωτών. 200 με 300 χιλιάδες παιδιά υπολογίζεται ότι εμπλέκονται σε ένοπλες συγκρούσεις. Η εκμετάλλευση των παιδιών στις ένοπλες ε, συγκρούσεις είναι κάτι το οποίο μας ε, σοκάρει ως κοινοβούλιο και επιπλέον να ακούμε δυσάρεστα νέα και από το Ιράν. Ανησυχούμε για την καταδίκη σε θάνατο